Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο κύριος Κορνιγέ και η κυρία Πατρίσια Λαλόντ πρόκειται να αντικαταστήσουν την κυρία Σιβλεγκουλάρ και την κυρία Ντεσσαρνέζ από τις 18 Πέμπτου του 2017. Λαμβάνει υπόψη ε, αυτόν τον ορισμό των γαλλικών αρχών το Κοινοβούλιο και θα τομοθετηθούν ως τακτικά μέλη με πλήρη δικαιώματα ε, στα όργανα